Ja, liebe Kolleginnen Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού και ε, χαίρομαι που ε, χαμογελάνε οι Γερμανοί γιατί χρησιμοποιώ τη γερμανική και όχι τη λατινική λέξη για τον τουρισμό και μπορεί νομίζω να γίνει και η, επό... η επίσημη μετάφραση στα γερμανικά ανάλογη. Λοιπόν, εάν δεν ε, υπάρχει καμία αντίρρηση νομίζω μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Τα πρακτικά, εάν ε, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση νομίζω μπορούν να εγκριθούν. Ωραία. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και αλλαγή του προϋπολογισμού. Οι συγητές είναι Σαγιάλα Σέντερ και Ντομινί Κρικέ. Δίνω τον λόγο στις δύο εισηγήτριες λοιπόν πρώτα απ' όλα. Ποια ξεκινάει. Κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ την συνεισηγήτρια Ινέες με την οποία δουλέψαμε και πολύ και καλά και τους σκιώδη συζητήσεις ταυτόχρονα, διότι όπως ξέρετε δεν είχαμε πολύ χρόνο να εργαστούμε. 15, οι τελευταίες 15 μέρες ήταν αργίες στην πράξη, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσουμε με όλους. Ωστόσο είχαμε μια καρποφόρα συνάντηση εργασίας με τους κύριους ηγητές που ευχαριστώ και γιατί ήταν παρόντες και γιατί ήταν δραστήριοι υπάκουοι και ταυτόχρονα παρέμειναν σε επαφή μαζί μας παρά το ότι είχαμε Πάσχα, διακοπές κλπ. Δεν ήταν βολική η περίοδος. Συνολικά υπήρχε μια αρκετά ευρεία συμφωνία, 15 συμβιβαστικά βασικές προτάσεις που υποστήριξαν πολλές ομάδες. Νομίζω ότι την έκθεση πρέπει να την παρουσιάσουμε σε δύο κομμάτια. Με τον κανόνα, με βάση το άρθρο 54, η Επιτροπή μας είναι ε, επί της ουσίας υπεύθυνη για το άρθρο 19 και 5.2α. Για τα άρθρα αυτά η δική μας επιτροπή έχει την βασική ευθύνη και ευτυχώς για τα άρθρα αυτά υπήρξε ομοφωνία. Το 19 ήταν αντικείμενος ε, πρότασης όλων των ομάδων για διαγραφή του συγκεκριμένου άρθρου και το 5.2α ήταν αντικείμενο και αυτό συνένεση. Η ιδέα μας ήταν να ξεκινήσουμε με ένα λεπτομερές αφροντίθετο από το πνεύμα του τσεχικής διοίκησης που ήταν να επανέλθουμε στην δουλειά που είχαμε κάνει μαζί πριν τα τελευταία δύο χρόνια λέγοντας ότι αυτό που έπρεπε να ληφθεί υπόψη πρέπει να γίνει με βάση τα κριτήρια και των guidelines και του μηχανισμού διασύνδεσης για την Ευρώπη για τα κύρια και τα επικουρικά δίκτυα. Ένα τομέα όπου καλύφθηκε εμπολής ε, από τις θέσεις μας. Ε, υπήρχε ομοφωνία στις προτάσεις αυτές. Δεν προτείναμε τροπολογίες για τα κεφάλαια 2, Β, Σ και Ε που στην ουσία είναι έργο της Ήτρε. Συμφωνήσαμε με τις, μεταξύ των δύο επιτροπών ένα είδος ε, συμφωνίας κυρίων όπου εμείς αλλάζουμε το κείμενο για εκεί που είμαστε η, επί της ουσίας υπεύθυνη επιτροπή και οι άλλοι κάνουν το ίδιο για το δικό τους τμήμα. Αυτό επιτρέπει να απλοποιήσουμε την ε, σχέση με την επιτροπή ΕΚΟΝ και beach που είναι υπεύθυνε για το θέμα και να λύσουμε το ζήτημα του άρθρου ε, του, της, ε, του επιμερισμού του άρθρου 54. Ω προς τα λοιπά είχαμε μια σειρά συζητήσεων, σημαντικές συζητήσει για το άρθρο 8 που δείχνει την προέλευση, που αναφέρεται στην προέλευση των πόρων. Ξέρετε ότι υπάρχει μια γενική υπεποίθηση στην Επιτροπή μας ότι δεν θέλουμε το Ταμείο Connecting Europe Facility και Ευρώπη 2020 να θυσιαστεί απευθείας σε μια πολιετή διαδικασία με στο Ταμείο Εγγύσεων του Μηχανισμού όλοι συμφωνούσαν ότι οι μη αναλωθέντες πόδι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα στην αιτήσια θέση του προπολογισμού. Αυτή ήταν και η θέση των επιτροπών. Μια δυσκολία είχε το εξή. Το ΕΛΚ πρότεινε πριν την αναθεώρηση του πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου να αναζητηθούν συμπληρωματικέ καλύψει από άλλα κεφάλαια του προπολογισμού. Δεν υιοθετήθηκε η πρόταση αυτή ωστόσο γιατί δεν, συμβα... δεν συμβαδίζει με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν έχει δηλαδή δημοσιονομική νομιμότητα. Αντίθετα, κάτι που εμπλούτησε την δουλειά μας είναι η πρότασή μας στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού προπολογισμού να ξανανοίξουν οι για την δυνατότητα να, να καλύψουμε τα κενά από άλλα κεφάλαια του προπολογισμού. Όλοι τους συμφωνούσαν για το θέμα αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να έρθουμε σε μια αιτήσια διαδικασία, τακτική αιτήσια διαδικασία του προπολογισμού, σεβόμενοι όσο περισσότερο γίνεται τα, τους πόρους αυτούς που εμπλουτίζονται από την νομοθετική διαδικασία και που είναι πόροι που είναι ήδη επιχειρησιακοί, λειτουργούν, βρίσκονται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού και κατά 95% έχουν αναλωθεί, κάτι που ε, επιτρέπει μια ορθή λειτουργία της, ε, του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ένα άλλο θέμα είναι το earmarking, ο τρόπο δηλαδή με τον οποίο και ε, οι πόροι και ο επαναπροσδιορισμός τους μπορεί να τεθεί σε συγκεκριμένα θέματα. Καταλάβουμε ότι ο καθένας είχε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και θέματα που ζητούσε, κάτι που οδήγησε σε ένα πολύ λεπτομερή κατάλογο τύπου μεταφοράς, περιβαλλοντικού θέματος, οριζόντιων ζητημάτων, μια πολύ περίπλοκη λίστα. Η θέση των συγητών ήταν να σταθούμε, να μείνουμε σε γενικές θέσεις, να μην να αποφασίσουμε ότι οι αναθέσεις θα γίνουν με βάση το πνεύμα των συζητήσεων στο Κοινοβούλιο και των προηγούμενων μηχανισμών. Δεν ε, θεωρήσαμε ωστόσο ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τις τροπολογίες για την επιμέρους ε, ανάθεση τοποθέτηση πόρων σε συγκεκριμένα θέματα. Όχι ότι δεν συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες των συναδέλφων που ήθελαν να υπογραμμιστεί η α ή β προσέγγιση ή τάση, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο, πολύ λεπτομεριακό, που εν τέλει ερχόταν και σε αντίθεση με το πνεύμα της απλοποίησης και της ταχύτητας που ε, περιγράφεται από τη διαδικασία αυτή. Υπογραμμίζουμε δε ταυτόχρονα και την ανάγκη να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί πολλές φορές. Είχαμε την ευκαιρία να, το, ε, να λάβουμε θέση και να ψηφίσουμε τα θέματα που θεωρούσαμε σημαντικά, διατηρώντας ε, υπόψη ότι η κοινοβουλευτική δουλειά που έχει γίνει έπρεπε να είναι ε, και για τις απευθείας και για τις έμεσες αναθέσεις. η αρχή των επιστροφών των, των, είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται ήδη και στο Συμβούλιο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δουλειάς που από κοινού κάναμε. Κλείνοντας πριν δώσω το λόγο στην Ινές, θέλω να πω ότι δεδομένη στις έντονης πίεσης που υπήρχε και θα υπάρχει προς το Κοινοβούλιο, διότι η θέση της Επιτροπής δεν είναι πολύ κοντά στη δική μας, άσε το Συμβούλιο, είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε μια εξαιρετικά μεγάλη ενότητα θέσεων ως Κοινοβούλιο. Οι συζητήσεις που θα γίνουν μετά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν θα είναι απλές. Όσο πιο δυνατή είναι η θέση μας, τόσο περισσότερα θα μπορέσουμε να περάσουμε. Αυτά εν ολίγης. Ευχαριστώ, είναι Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντομινίκ Ρικέ Κάναμε μια καλή δουλειά, συνέχεια ίσως αυτών που είχαμε κάνει στο παρελθόν να ευχαριστήσω ιδίω όλους τους συναδέλφους και τους σκιώδης ηγητέ και τους υπόλοιπου συναδέλφου που παρουσίασαν τροπολογίες και για το ότι έδειξαν τη γενεοδορία να δεχθούν σε κάποιε περιπτώσεις να θυσιάσουμε εν μέρη το κείμενο των τροπολογιών τους, ελπίζοντας όχι όμως το πνεύμα τους προς όφελος ε, στέρεων συμβιβαστικών λύσεων που διατηρούν αυτή τη σημαντική ενότητα με βάση την οποία η Επιτροπή μας ήδη από τον κανονισμό ΤΕΝ είχαμε κατορθώσει να πετύχουμε πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι και στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα που έχουμε να κρατήσουμε μία στεναρή ενωτική θέση αποτελεί τμήμα της επιτυχίας και ταυτόχρονα της ταχείας κινητοποίησής μας κατά του προϋπολογισμού ε, κατά της ε, αποδυνάμωσης του προπολογισμού Juncker εις βάρος έργων που εμείς έχουμε προωθήσει όπως το Connecting Europe Facility αλλά και την αναγκαιότητα να είμαστε προσεκτικοί διότι όπως είπε ο Ντομινίκ νωρίτερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έξω από το Κοινοβούλιο ανεβαίνει, αυξάνεται το λόμπι εις βάρος μας πιέζοντας ή τέλο πάντων κατηγορώντας μας ότι θέλουμε να μπλοκάρουμε ή και να αποτρέψουμε το σχέδιο Γιούνκερ, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να φροντίσουμε με κάθε τρόπο να συμπληρώσουμε αυτό που ήδη έχει υλοποιηθεί με το υπολογισμό της Ένωσης, προσθέτοντας και αυτήν την αρχή της προσθετικότητας μια σειρά νέων πόρων στον προπολογισμό, που ή δεν χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται σε stand-by αυτή τη στιγμή και που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για, την, για το Ταμείο Εγγύησεων. Είναι σημαντικό λοιπόν η δουλειά που κάναμε για να έχουμε κοινή θέση ε, να πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους σας για την κατανόηση που δείξετε στο ότι δεν πήγαμε παραπέρα, δεν ανοίξαμε άλλα κεφάλαια του προπολογισμού που επέτρεπαν, τον είχαν μια σχέση με την γενική θέση του Κοινοβουλίου, εν μέρει ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν για να ασκηθεί πίεση, αλλά προς το παρόν ε, τη στιγμή της ψηφοφορίας πρέπει να είναι σαφές ότι εμείς δεν μπλοκάρουμε το σχέδιο Juncker, αλλά ζητούμε πόρους ε, που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τα, σχέδια, για τα έργα αυτά. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους για την ικανότητα γεωγραφικής διαφοροποίησης και τομεακής διαφοροποίησης των έργων που μπορούν να ληφθούν υπόψη, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κερδίζουν μόνο μία-δύο χώρες από το σχέδιο Γιούγκερ αλλά ότι θα υπάρχει δυνατότητα να μετάσχουν όλοι, να μπορούν να, να μετέχουν σε αυτό. Για τις επιστροφές τώρα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των επιστροφών, των ειδικών επιστροφών για συγκεκριμένα θέματα, για συγκεκριμένους τομείς που γνωρίζει η Επιτροπή μας, ε, φερειπίν ε, επιδοτήσει ιδεοδρόμων, αλλά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επανέλθουν στον γενικό προπολογισμό, εξασφαλίζοντας την διατήρηση της εγγύησης, κάτι που όμως δεν θα πρέπει να, εμποδίζει ό,τι επενδύουμε ή ό,τι επενδυθεί στο μέλλον να τηρεί αυστηρά τις προϋποθέσεις των κανονισμών TEN διευρωπαϊκών δικτύων και Connecting Europe Facility και για το σιδηρόδρομο αλλά και ταυτόχρονα και άλλες πρωτοβουλίες το urban mobility, την προσβασιμότητα, μια σειρά δηλαδή νέων ε, πρωτοβουλειών που θα δώσουν τη θέμενη αξία τα διάφορα έργα των μεταφορών. Τελειώνοντας, ευχαριστώ γιατί σε κάποια από τα έργα που υποβλήθηκαν από κάποιες ομάδες για να διευρυνθεί ή για να ανοίξουμε τον κατάλογο των έργων που υιοθετήσαμε στους δύο προγενέστερους κανονισμούς, για μένα τουλάχιστον θα προτιμούσα κάποια από τα έργα που αφορούν την περιοχή μου ε, να μην αναφέρονται στο σχέδιο Γιονγκέν, Να σας πω γιατί. Γιατί στο σχέδιο, το σχέδιο Γιονγκέν είναι ένα σχέδιο για έργα που έχουν μεγάλο κίνδυνο, που περιέχουν μεγάλο κίνδυνο και η βιωσιμότητα των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε μακρύ χρονικό ορίζοντα. Άρα πρέπει να βγει στην αγορά. Άλλα μικρά σχέδια, το missing links, τον, ε, τα διασυνοριακά missing links δεν χρειάζονται κάτι τέτοιο, χρειάζονται άμεσες ενισχύσεις με σωστή στοχοθέτηση που εξαρτώνται περισσότερο από την λογική του Connecting Europe Facility ή των διευρωπαϊκών δικτύων και όχι τόσο του σχεδίου Juncker που τέλος πάντων θα πάει στις τράπεζες και θα δούμε τι θα βγάλει. Αυτά τα ολίγα. Ευχαριστώ. Η γραμμή ωστόσο Μικάμ Φρανέρων καλύτερα να περάσει μέσω των εθνικών επιδοτήσεων και όχι μέσω του σχεδίου Γιονκέρ. Ευχαριστώ ο Μάρκος Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά θα θέλαμε σε κάποια πράγματα πιο σαφείς ε, διατυπώσεις σε σχέση με την εναλλακτική της ε, χρηματοδότησης, αλλά εγώ είμαι δημοκράτης και βεβαίω. Ε, μπορώ να αποδεχτώ τις πλειοψηφίες που υπάρχουν στην Επιτροπή και άρα δεν είναι δυνατόν ευθύς ε, εξ αρχής ε, να χρησιμοποιήσουμε λεφτά από το αποθεματικό. Είναι κρίμα. Εγώ επαναλαμβάνω το ότι καμία χώρα δεν θα το πρόσεχε. Είχαμε βρει τις δυνατότητες να διατηρήσουμε την εθνική κατανομή που υπήρχε. Παρόλα αυτά, ε, βεβαίως θα υποταχθούμε στη τη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή, αλλά Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση θα υπάρχει δυνατότητα και σας ευχαριστώ και για αυτή την παραχώρηση. Η δυνατότητα λοιπόν να εξετάσουμε όλες τις γραμμές ε, του προϋπολογισμού ε, για να δούμε αν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ξανά το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. αλλά αυτό ο συμβασμός είναι κάπως ε, επικίνδυνος γιατί θα μπορούσε να επιβαρύνει νομίζω την κατάσταση και θα ήθελα άρα να μπει εδώ πέρα πως ναι θέλουμε αυτή την επανεξέταση αλλά δεν θέλουμε οι χώρες της συνοχής ή οι ασθενέστερες χώρες να υποφέρουν από αυτό. Θα προτείνω μια διατύπωση το απόγευμα προς αυτή την ε, κατεύθυνση Το ένα είναι αυτό. Δεύτερο που θα θέλαμε να αλλάξει και το είπαμε στο συμβαστική πρόταση 8.2 είναι ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε μόνο αυτή την δυνατότητα αλλά θέλουμε από την Κομισιόν μια δεσμευτική συμφωνία. Να τους πούμε δηλαδή πρέπει στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση να τα ξαναδείτε όλα αυτά. Όχι μπορείτε άμα θέλετε κτλ. Δεσμευτική συμφωνία. Αυτό βεβαίω σε σχέση με το δίκτυο ασφαλείας που λέγαμε για τις χώρες ε, συνοχής νομίζω θα βρει μια πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Αυτά τα δύο ήθελα να πω για το 8.2 τη συμβιβαστική πρόταση. Συμφωνούμε και με την γεωγραφική ισορροπία γιατί βέβαια ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται πάλι με την στάθμιση των ε, ασθενέστερων περιοχών. Γιατί τα δισεκατομμύρια τα οποία φεύγουν από το μέσο ενδιόντα της Ευρώπης δεν φεύγουν από τις ασθενέστερες χώρες αλλά από τις υπόλοιπες και πάνε ως εγγυήσεις. Και να πούμε τώρα ότι θέλουμε τα έργα να επικεντρωθούν στις χώρες της συνοχής, τις ασθενέστερες δηλαδή, σημαίνει ε, τις προστατέψαμε μία φορά τις χώρες της συνοχής με τα 11 δις και τώρα παίρνουν και τα 3 δισεκατομμύρια επιπλέον. Κάπως υπερβολικό. Παρακαλώ να είμαστε κάπως δίκαιοι ο ένας ε, με τον άλλον. Εμείς επιδείξαμε ένα συμβιβαστικό πνεύμα και το ίδιο αναμένουμε τώρα και από τους άλλους. Και κάτι άλλο βεβαίω, το οποίο δεν νομίζω να συμφωνήσουμε τόσο εύκολα στο τέλος, είναι οι όροι με τους οποίους ε, γίνεται ακριβώ ε, η ενίσχυση αυτή με όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία πάνε κάπως προς μια κοινωνική κατεύθυνση. Δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό με ε, την καινοτομία, τις μικρομισές επιχειρήσεις, τις υποδομές. Οπότε, εδώ πέρα πραγματικά θέτουμε σε κίνδυνο το σχέδιο Juncker. Γι' αυτό εμείς ως ΕΛΚ θεωρούμε σαφώς ε, πως ε, στη συμβαστική αυτή πρόταση μια στιγμή που ποιο νούμερο είναι το 5 νομίζω ναι συμβαστική 5 ε, σας παρακαλώ να το ξαναδούμε απόψε γιατί εμείς θεωρούμε πως κάπως παραπάει. Γιατί μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το σχέδιο Γιούνκερ και δεν θα μπορέσουμε να το δεχτούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Να πετύχουμε μια συμφωνία. Τώρα, άμα δει κανείς τη σούμα, Ακούγονται κάπως δραματικά τα πράγματα. Μιλάμε για 20 συμβαστικέ, τις οποίες μπορούμε να δεχτούμε όμως και δύο σημεία έχουν μείνει ανοιχτά, στα οποία είπα πως θέλουμε κάποιες αλλαγές και καλό θα ήταν να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε. Και βεβαίω όσο πιο ενωμένοι είμαστε, όσο πιο μεγάλη βαρύτητα θα έχει η θέση μας μετά. Ρόμπερτ Σίλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ευχαριστώντα τους δύο συνεισηγητές. Ήταν νομίζω καλή επιλογή και οι δύο τους, ε, γιατί είχαν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και στο παρελθόν. κατάσταση είναι ανησυχητική. Πρέπει να το πω εξ αρχής και το κυριότερο που με ανησυχεί είναι αυτή η αλλαγή που γίνεται στις πηγές χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ κύριε Πίπερ για αυτά που είπατε. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι σημαντικό να ξαναδούμε στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ε, αναθεώρηση του προϋπολογισμού άλλες πηγές, χρηματοδότηση από άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού. Όμως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και δυσκολίες στην μεσοπρόθεσμη ε, αναθεώρηση. Έχουμε υποστηρίξει και θα υποστηρίξουμε μάλλον τις προτάσεις που αναφέρονται στους σιδηροδρόμους και πρέπει να ε, τονίσουμε τη σημασία της γεωγραφικής ουδετερότητας το είπε ο κ. Πίπερ ότι υπάρχει ήδη αυτό σήμερα. Γιατί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων απευθύνεται και αφορά και χώρες που δεν είναι χώρες συνοχής. Αυτή τη στιγμή οι χώρες αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων. Και δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτό το νέο ταμείο. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε έτσι ώστε να μην υπάρξουν ανισότητες στη γεωγραφική κατανομή των πόρων. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την κατανομή των πόρων κατά κλάδο. Δεν θα θέλαμε να υπάρξει ξαφνικά ε, μια μετακίνηση χρηματοδοτήσεων, χρηματοδότησης προς την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων για παράδειγμα. Έχω 20 χρόνια στην πολιτική και δεν θα έλεγα ότι είμαι αφελής. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να κάνουν επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις. Και αυτές έχουν βασιστεί σε πόρους earmarked. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, δεν υπήρχε καμία διάθεση στι χώρε αυτέ να γίνουν επενδύσει σε άλλε χώρε, σε τρίτε χώρε, σε αλλα άλλα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι όσο πιο ανοιχτά συζητούμε μεταξύ μα τα θέματα, τόσο καλύτερα καταλήγουμε σε συμβιβαστικέ θέσεις, σε κοινέ θέσεις. Πάντως, α μην περιμένουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα τη συμφωνία θα είναι εύκολη. Ευχαριστώ, Μαρία Κίλε μου. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvin lyhyesti haluaisin kiittää. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνηθιγητές για το εξαιρετικό έργο τους, ιδιαίτερα δεδομένων των δυσκολιών που είχαν να αντιμετωπίσουν με τις αργίες κτλ. γιατί όλοι προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας με αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και κανείς νομίζω δεν γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει ακόμα. Με ανησυχεί λίγο αυτή η τάση που διαβλέπω να ξαναανακαλύπτουμε τον τροχό στην στα χρηματοδοτικά μέσα, στους πόρους χρηματοδότηση, τη διάφορα ταμεία, χωρίς κανείς στην πραγματικότητα να απαντά στο βασικό ερώτημα πού θα βρούμε τα χρήματα μήπως θα ήταν καλύτερα να αξιοποιούμε ε, με βέλτιστο τρόπο τα ήδη υπάρχοντα ταμεία και τα φυστάμενα χρήματα. Ευχαριστώ, Καρίμα Δελή. Euh, Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν. Το πρόγραμμα Juncker πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα έξυπνης ανάκαμψης που πρέπει να λάβει υπόψη και το μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι έξυπνη. Οι μεταφορές θα πρέπει στο μέλλον να λάβουν υπόψη το φαινόμενο της αλλαγής του κλίματος, το περιβάλλον, τις ανάγκες σε ενέργεια. Άρα η πραγματική, αυτό που πρέπει να πούμε για το πρόγραμμα Juncker είναι σε τι θα χρησιμεύσουν οι επενδύσεις στις μεταφορές. Ευχαριστώ για τις συμβαστικές προτάσεις. Εμείς οι οικολόγοι συμφωνούμε με πολλές από τις συμβαστικές προτάσεις με την εξαίρεση του πιο σημαντικού, του άρθρου 5 δηλαδή, όπου ε, σημειώσετε τις ε, θέσεις των οικολόγων στη συμβαστική πρόταση, αλλά δεν τις λάβατε υπόψη τουλάχιστον τις βασικές μας θέσεις. Εμείς είχαμε πει, για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε 60% των επενδύσεων κατελάχιστον να πάνε στις ιδεοδικέ μεταφορές. Να προσανατολίσουμε 10% των επενδύσεων για να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα με το ποδήλατο, με το περπάτημα. Που Πουθενά να είναι αυτά για το σχέδιο Γιούνκερ είπαμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ε, ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών. Δεν υπάρχει στο πέντε αυτό. Πολλά πράγματα δεν υπάρχουν. Η βούληση να ενισχύσουμε αστική, βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Το θέμα του θορύβου. Ούτε καν το φύγουμε. Αυτά είναι θέματα καυτά σήμερα. Το κόστος και είναι κρίσιμο γιατί αν από το ξεκίνημα δεν ξέρουμε που πάμε, δεν θα προχωρήσουμε με έξυπνο τρόπο. Αν έχουμε σαφείς στόχους, σαφή, σαφή ορόσημα, και στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα της τοπικής κοινωνίας, τι θα κάνουμε. Σήμερα πρέπει να προσανατολίσουμε σωστότερα το κείμενό σας. Ξέρω ότι αύριο ψηφίζουμε, μπορεί να βρεθούμε στο περιθώριο, αυτά ήθελα να σας πω ως οικολόγος πάντως. Στο D'Amato. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους εισηγητές. Εν γέννη είμαστε ικανοποιημένοι. Εκτιμήσαμε την βούληση επίτευξης συμφωνίας και την ανάδειξη της σημασίας των μεταφορών και στο σχέδιο Juncker και στην Ευρώπη. Μία παρατήρηση μόνο για να σταθώ σε ένα θέμα. την δυνατότητα που αφήνεται να εμπλακεί και το CF. Εμείς θα προτιμούσαμε με τη διαγραφή του 19 να... Αλλά δεν μπορούμε, εμείς προτιμούμε τη διαγραφή του 19, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό πρέπει να μπει, αυτή η δυνατότητα μπορεί να μπει στα εκτιμώντας, έστω και σαν και όχι ως προτεραιότητα. Το υπογραμμίζω αυτό, θα ήθελα και στην, ε, στην σκέψη να φύγει η μνήμη αυτή. Στο Κριστίν Ρεβόνταλο. Merci, Président. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές για το δύσκολο έργο τους δεδομένες της ποσότητας, του αριθμού των ε, τροπολογιών που είχαν υποβληθεί, όπως έλεγε και η Νέσ πριν από λίγο. Όλοι, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουν να δουν αυτή την ε, ανάκαμψη της οικονομίας και της ανάπτυξης. Γι' αυτό νομίζω προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σχέδιο Juncker έτσι ώστε να είναι πραγματικά προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό προσπάθησα να κάνω και εγώ με τις τροπολογίες που υπέβαλα και σας ευχαριστώ που τις λάβατε υπόψη σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο, έτσι ώστε το σχέδιο Juncker να μπορέσει να βοηθήσει όλες τις χώρες θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του ελλείμματος, για παράδειγμα είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, είναι θεμελιώδους σημασία και πιστεύω είναι ε, η τελευταία φορά, είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είχε πει και ο Πρόεδρός της, να ανταποκριθεί στις απαιτήσει και στις ε, προσδοκίες των πολιτών. Δεύτερον, είναι σημαντικό να θεωρήσουμε ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να εξυπηρετήσει την αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, ε, λαών και κρατών. Ακόμα περισσότερο χρειάζεται αυτή η ελληνική τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει το σχέδιο και να βοηθήσει κατά κύριο λόγο τις χώρες εκείνες που έχουν πληγεί ε, σε μεγάλο βαθμό από την κρίση. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για τον προϋπολογισμό δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι η Κομισιόν ανησυχεί από την προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Δεν είναι ότι δεν μας αρέσει το μέσο αυτό. Μας αρέσει και γνωρίζουμε πως η πρόταση δημιουργεί δυσκολίες, αλλά είμαστε πεπισμένοι πως όταν προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικέ είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν όχι αδύνατον, να βρεθούν αυτές. Ε, πρέπει να λειτουργήσουμε υπό τον τίτλο 1α του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και όταν γίνεται αυτό έχουμε επιλογή μεταξύ μικρών περικοπών σε μεγάλα προγράμματα ή το αντίστροφο. Οπότε προτιμούμε τις μικρές περικοπές σε μεγάλα προγράμματα για το θέμα της ευελιξίας. Θέλω εδώ να επιμείνω στο εξής. Είναι δύσκολο να βρούμε 350 δισεκατομμύρια για επενδύσεις με 21 δισεκατομμύρια δημόσιο χρήμα εάν δεν έχουμε μέγιστη ευελιξία. Οπότε η όλη αυτή η ιδέα γεωγραφικής ή τομεακής κατανομής στην πράξη θα δημιουργήσει πρόβλημα για να πετύχουμε τον στόχο αυτό των 315 δισεκατομμυρίων. Πρέπει να αντιληφθείτε πως υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη και του ΕΤΣΕ. Στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη εξοδεύουμε δικά μας λεφτά και μπορούμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσουμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρεια το τι θα κάνουμε. Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις δημόσιες δαπάνε, αλλά να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια με όσο το δυνατόν λιγότερα δημόσια. Οπότε, όσο πιο πολλού όρου βάζουμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να προσελκύσουμε δημόσιες επενδύσεις. Υπό το πρίσμα αυτό όλες αυτές οι ιδέες για ε, λεπτομερείς απαιτήσει ή γεωγραφική κατανομή θα μπορούσαν να αποδεχτούν προβληματικές. Για το θέμα της συνοχής καταλήξαμε πάρα πολύ γρήγορα στο συμπέρασμα πως εάν έχουμε γεωγραφικό φάκελο μπορούμε να είμαστε τελικά αυτό να αποδεχθεί κατά των συμφερόντων των χωρών της συνοχής. Στη φιλοσοφία του ταμείου αυτού πρέπει να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές σε έργα που επιλέγονται με βάση την αξία τους. Εάν έχουμε γεωγραφική κατανομή, δημιουργούμε μια υποψία για το σκεπτικό του κάθε έργου και άρα αμφιβολία στον ιδιώτη επενδυτή για το γιατί ακριβώς λάβαμε την απόφαση να υπάρχει εγγύηση σε ένα έργο. Μισθέμε το έργο να μπορεί να ανταγωνιστεί επίσης όρις, γι' αυτό ακριβώς αυξάνουμε την τεχνική αρρωγή, οπότε όλοι ανεξαρτήτως της χώρας μπορούν να υποβάλουν έργα υψηλή ποιότητας χωρίς κάποια πρώτερη κατανομή. Τούτου λεχθέντος. Η Κομισιόν προσπάθησε πάρα πολύ να προστατεύσει τις χώρες συνοχής, δεν προτείναμε περικοπές σε διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία συνοχής και όσον αφορά το μέσο συνδέοντα την Ευρώπη προσπαθήσαμε ακριβώς να προστατεύσουμε τις χώρες συνοχής και καταλαβαίνουμε πως εάν πρέπει να γίνουν προσπάθειες ε, στην αναθεώρηση θα πρέπει να δούμε και τις χώρες συνοχής. Αυτά από μένα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η Νέσα Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Δεν κατάλαβα βέβαια καλά σε κάποιες περιπτώσεις ποιο ήταν το πρόβλημα. Ο κύριος Πίπερ αναφέρθηκε σε δύο θέματα που δεν τα κατάλαβα. Πρώτον, τις χώρες συνοχής. Νομίζω ότι το συμβαστικό κείμενο έλεγε ότι δια, διασφαλίσαμε μια ε, γεωγραφική διαφοροποίηση του αντικτύπου του ταμείου αυτού, ώστε να μην επικεντρώνεται η δύναμη του μέσου αυτού σε μία-δυο χώρες γιατί πάντα λέγαμε για κάποια μεγάλα έργα που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες στις συνοχές θα προστατευτούν. Προστατεύονται. Ε, Εφαρμόζεται ο κανονισμός, είναι αυτές που είναι και φροντίζουμε να μπορούν τα νέα τα κράτη συνοχής που βοήθησαν πολύ στην διαμόρφωση του Ταμείου με, τον, με τα 11 δις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το ξεκίνημα του εργαλείου αυτού στα πρώτα χρόνια της εγγύησης κυρίως να υφίστανται αλλά με πολύ πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προπολογισμό από ό,τι μέχρι τώρα. Δηλαδή ό,τι δεν χρησιμοποιείται επιστρέφεται στα κράτη-μέλη ενώ έχει προπολογιστεί. Εάν ο προπολογισμό είναι επαρκή, το κοινοβούλιο όπω έχουμε ζητήσει πρέπει να μπορεί να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό χρησιμοποιεί για ευρωπαϊκά έργα. Αυτό. Μετά, μίλησε για το συμβασμό 5, ότι υπήρχε ένα πλεόνασμα στα κοινωνικά θέματα. Εγώ το κοιτάω, το ξανακοιτάω, δεν βλέπω ούτε μία μνήα. Μία από τις υποχρεώσεις του σχεδίου Γιούνκερ είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα των χωρών του Νότου. Δείτε κύριε Πίπερ και εσείς την χώρα σας όπου πρέπει να ενισχυθεί για παράδειγμα και η ποιότητα της δουλειάς, ακόμα και στη δική σας χώρα. Τα υπόλοιπα είναι επενδύσεις σε ανταγωνιστικότητα, γίνεται λόγος. Το πρώτο θέμα όλων είναι ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία με την στρατηγική Ευρώπη 2020, μια στρατηγική καινοτομίας κατά βάση και σχέσεων με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, όχι αποκλειστικά με τα κοινωνικά θέματα, την απασχόληση. Τέλο δεν καταλαβαίνω τι ανησυχεί, Αν μπορεί να μου έφυγε κιόλας, οπότε δεν μπορεί να μου το εξηγήσει. Τώρα, καταλαβαίνω τις ανησυχίες των συναδέλφων για το ότι οι στόχοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους στόχους που έχουμε θέσει και όχι για την οικοδόμηση, ας πούμε, την, την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Ε, η άποψή μας είναι ωστόσο ως επιτροπή ότι όλα τα έργα που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα Juncker να γίνονται με βάση τις ε, βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, τον κανονισμό TEN και τον κανονισμό Connecting Europe Facility. Οι αξίες δηλαδή να μπορούν να ε, πηγαίνουν κατά βάση στο σιδηρόδρομο με συνέργεια στο urban mobility, μια πιο βιώσιμη ε, μορφή μεταφορών, πιο πράσινη μορφή μεταφορών. Δεν χρειάζεται να το λέμε και να το ξαναλέμε όμως. Από το ξεκίνημα εμείς είπαμε ότι όλα είναι μέσα στα πλαίσια του Connecting Europe Facility και των TEN εν γέννη. Το earmarking του 60% για τον ε, για το σιδηρόδρομο, εντάξει καλό χρυσό, αλλά δεν δίνει ευελιξία σε ένα ταμείο που δίνει φιλανθρωπικές βοήθειες στην ε, μορφή μεταφοράς που θέλουμε, αλλά για να επιτρέψουμε στα επενδυτικά ταμεία τα ιδιωτικά να καταλάβουν ότι τα έργα αυτά είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά βιώσιμα. Αυτός δηλαδή που θα δανείσει να ξέρει ότι θα πάρει πίσω κάτι. Αλλιώς ε, δεν μπορούμε να μιλάμε για συνεχείς επιδοτήσεις ας πούμε του τρένου, του θορύβου κλπ. Το σχέδιο γιούνκερ είναι κάτι παραπέρα. Μην φτάσουμε σε χειρότερη κατάσταση. Βασικές αρχές λοιπόν του CF και του TEN, αλλά ταυτόχρονα δείχνοντας τις καθοδητήριες γραμμές που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Για την κυρία Κιλόνεν μιλάμε για, τα υφιστάμενα, για τους υφιστάμενους πόρους. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό. Εγώ λέω να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότητα αυτά που έχουμε. Δεν ζητάμε ούτε φράγκο παραπάνω. Ζητάμε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που δαπανάται κακά μέχρι τώρα διότι επιστρέφονται κονδύλια ανακτώνται δηλαδή πόροι που δεν δαπανώνται και επανέρχονται στα κράτη-μέλη. Μιλάμε για ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όχι εθνικό. Αυτό που θέλουμε είναι να χρησιμοποιείται καλύτερα ούτω ώστε το σχέδιο Γιούνκερ που θέλει να δημιουργήσει πλούτο ε, απασχόληση σε μια ευρωπαϊκή δυναμική να χρησιμοποιείται καλύτερα, αποτελεσματικότερα. Για τις προτάσεις που γίνονται, σας θυμίζω συνάδελφοι, ότι πρέπει να κάνουμε ένα mainstream με τις γενικές προτάσεις του Κοινοβουλίου. Τις ΣΥΤΡΕ, κυρίως δε, των επιτροπών προϋπολογισμού, ελέγχου του ε, προϋπολογισμού, συγγνώμη, και της Οικονομικής Επιτροπής. Να βρούμε λοιπόν μια διατύπωση που είναι όσο πιο κοντά στο mainstream που χρειάζεται το Κοινοβούλιο για να βγάλει μια πλειοψηφική θέση. Όπως σας θυμίζουμε, μας πιέζουν οι πάντες, κομισιόν, κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη πολίτες θεωρούν ότι εμείς κλωτσάμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία για να καταστήσουμε σαφές ότι το Κοινοβούλιο θέλει αποτελεσματικότερο ταμείο στα πλαίσια ιδίως των υποδομών μεταφορών που θα χρησιμοποιείται σε συμφωνία με τις αρχές και τις αξίες που έχουμε, που διαθέτουμε και που επιτρέπουν να δημιουργηθούν νέα βιώσιμα έργα για τα οποία οι δημόσιοι πόροι δεν είναι παρικοί και άρα χρειάζεται η εμπλοκή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχει να δαπανίσει και που τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να ε, επενδύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή τους συναδέλφους. Το πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι με αυτόν τον κανονισμό τώρα δεν προσπαθούμε να ξαναγράψουμε από την αρχή πολλούς και διάφορους άλλους παλαιότερους κανονισμούς. Υπάρχει το CEF, υπάρχει το Connecting Europe, υπάρχει το ε, δεν ε, υπάρχει το δημοσιονομικός κανονισμός και δεν προσπαθούμε τώρα να τους αλλάξουμε όλους αυτούς. Αντιθέτως, το σημαντικό είναι να καταφέρει το Κοινοβούλιο να συντονίσει τη θέση των τεσσάρων αρμόδιων επιτροπών του η οποία κάθε μια φυσικά έχει την τάση να εκφράζει τις θέσεις που είναι πιο κοντά στο δικό της αντικείμενο, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε ε, υπερβολική απομάκρυνση από το, το πλαίσιο του κανονισμού αυτού. Πρέπει να παραμείνουμε στο πλαίσιο του κανονισμού. Σημείωσα λοιπόν όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι και ε, η ομιλία του Μάρκου με παρεκκρέντωσε λίγο γιατί έλεγε μία θέση και αμέσω μετά την αντίθετη. Χρειάζεται λοιπόν, λέμε, να προχωρήσουμε γρήγορα με την υλοποίηση των διαφόρων σχεδίων αλλά ταυτόχρονα να ε, προστατεύσουμε τις χώρες της συνοχής αλλά αμέσω μετά μα λέει ότι ακριβώ εκείνα τα σχέδια τα οποία τον προβληματίζουν είναι εκείνα που θα υλοποιηθούν στα κράτη-μέλη τη συνοχή. Δεν κατάλαβα λοιπόν ακριβώ ποιο ήταν το αντικείμενο τη παρέμβαση του. Αυτό που είναι ξεκάθαρο και το λέω και για τον Ρόμπερτ. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν θα μεταβληθεί κατά τρόπο ε, σημαντικό. Υπάρχουν κάποια μικρά κονδύλια τα οποία περισσεύουν, για αυτά συζητούμε. Υπάρχουν λοιπόν οι χώρες που υποφελούνται από το Ταμείο Συνοχής. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες χώρες οι οποίες είναι σε ε, ε, ε, κατάσταση δύσκολη χωρίς να υποφελούνται από το Ταμείο Συνοχής. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τα κράτη συνοχής είναι τα πιο επισφαλή. και δεν πρόκειται να αλλάξει η κατανομή των κονδυλίων αυτών στον το, ταμείο συνοχή στο πλαίσιο του πολιετού δημοσιονομικού σχεδίου. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να πάμε πιο πέρα, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρχει αξιοποίηση των επιπλέον κονδυλίων. Επομένως, ε, δεν μιλούμε ούτε τώρα, ούτε με την αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής. Επομένως, οι ανησυχίες που εκφράστηκαν θα έλεγα ότι έχουν βρει την απάντησή τους. Είναι άνευ αντικειμένου δεν πρόκειται να υπάρξουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Καρίμα, καταλαβαίνω τι λέτε. Αναφέρατε μια σειρά ζητημάτων τα οποία οι οικολόγοι είχαν θίξει. Αλλά εδώ δεν προσπαθούμε να επαναλάβουμε το κείμενο της, ε, του Connecting Europe Facility. Έτσι κι αλλιώς το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη είναι αυτό που δίνει την πολιτική κατεύθυνση και για τα επιπλέον σχέδια που θα χρηματοδοτήσουμε με το σχέδιο Juncker. Επομένω δεν έχει νόημα να, αρχίσουμε να αναφέρουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση του ποδηλάτου, το α ή το β ζήτημα. Οι συνεισηγητές το έχουν καλύψει αυτό με μια παραπομπή στο Connecting Europe Facility. Επομένως, αν και αντιλαμβάνομαι τις, τις ανησυχίε σας και τις θέσεις σας, πρέπει να φροντίσουμε ο μηχανισμός αυτός που είναι εγκυοδοτικός μηχανισμός θα έχει την ευελιξία που του χρειάζεται και θα προχωρήσει όσο γρήγορα χρειάζεται. Υπάρχουν οι υπόλοιποι κανονισμοί, υπάρχει το Common Acting Europe Facility, υπάρχει ο κανονισμός για τα ταμεία συνοχής και αυτά αρκούν για τα υπόλοιπα θέματα που έδειξαν οι συνάδελφοι. Και γι' αυτό έχουμε ε, εντάξει και στο κείμενό μας τις παραπομπές στα υφιστάμενους κανονισμούς. Για να καθοδηγήσουμε και την υλοποίηση ε, της απόφασης αυτής από την Επιτροπή στο μέλλον. πριν γίνει η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορούμε να το αποσταθεροποιήσουμε αυτή τη στιγμή τον προϋπολογισμό της Ένωσης δίνεται η δυνατότητα μέσω των συνδικών της Ένωσης να υιοθετούνται τέτοια μέτρα εγγυοδοτικά, δημιουργία ταμείων εγγύησης και αυτό το ταμείο των 8 δισεκατομμυρίων είναι ένα τέτοιο ταμείο αλλά υπάρχει και η ε, απέτηση να υπάρχει η δημοσιονομική ασφάλεια και γι' αυτό κάνουμε την αναφορά στις επιστροφές του προϋπολογισμού για να υπάρχει μια κάποια ασφάλεια για το πού θα βρεθούν τα απαιτούμενα χρήματα. έλεγα ότι αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες των διαφορών συναδέλφων, αλλά θα έλεγα ότι το κείμενο στο οποίο έχουμε καταλήξει τις καλύπτει, γιατί ταυτόχρονα προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και να εξασφαλίσουμε και την ευελιξία που χρειάζεται και την παροχή βοήθειας στις χώρες που την έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, οι οποίες δεν είναι πάντα οι χώρες συνοχής. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, γιατί αυτό που είπε είναι πραγματικά θεμελιώδης σημασία και συμφωνώ μου μας θυμήσατε ότι το ε, σχέδιο Juncker και το ΕΤΣΕΠ είναι ε, το, το, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι δύο διαφορετικοί μηχανισμοί, διαφορετικής φύσεως μηχανισμοί. Άλλο πράγμα είναι η επιδότηση, άλλο πράγμα είναι η γης. Είναι διαφορετικό ειδών πολιτικές και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα που προσφέρονται να αντιμετωπιστούν καλύτερα με εγγυήσεις, με εγκυοδοσία, με επιδοτήσεις, ούτε το αντίστροφο. Όπως ε, είπατε, σωστά δεν πρόκειται να, να, αγγίξουμε τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί ούτε για τα Ταμεία Συνοχής, ούτε για την ΚΑΠ, ούτε για τα μεγάλα, άλλα μεγάλα ε, προγράμματα. Φαίνεται λοιπόν ότι η Επιτροπή θα εμείνει στη θέση της, όπως σκοπεύει να εμείνει και στη δικιά του, η οποία ευελπιστώ να είναι και πολύ ξεκάθαρη. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μακρά και δύσκολη συζήτηση μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο εισηγητές. Η ψηφοφορία είναι αύριο στην Επιτροπή μας και την εβδομάδα της, ε, τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου στην Ολομέλεια. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάθεξης. την διαδικασία για τις ακροάσεις των επιτρόπων διδάγματα από τη διαδικασία του 2014. Ε, εγώ είμαι ο εισηγητής. Σήμερα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Αύριο το πρωί έχουμε ψηφοφορία. Έχω γράψει και μία επιστολή. Συνολικά έχουμε 19 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Έχω υποβάλει κάποιες συμβαστικές ε, για τις ε, παραγράφους 1 και 2 που περιέχουν όλη την ουσία. Μια προφορική τροπολογία για την παράγραφο 3 μαζί με τον Βιμ Φαντεκάντ. επίσης θα ε, σας προταθεί και βεβαίως Θα δούμε τι θα γίνει με την διαδικασία η οποία οδήγησε στον ε, ορισμό του ε, Επιτρόπου Μεταφορών. Είχαμε επίση και την αξιολόγηση της διαδικασίας από την κυρία Βιολέτα Βούλτς. Υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες που δεν καλύπτονται από αυτές τις συμβαστικές προτάσεις και άρα θα ψηφιστούν ξεχωριστά. Θα δώσω τώρα τον λόγο στους και όδης Ο Βίμφαντε Κάμπ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, ο συντονιστής μας ακόμα ταξιδεύει. Εξ του ΕΛΚ να πω πως δεν έχουμε κάποια προβλήματα με τον συμβιβασμό αυτό και τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Πάρα πολύ απλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σμαήλ Ερτού. Ευχαριστώ και εμείς ε, σοσιαλιστές μπορούμε να πούμε πως ε, συμφωνούμε εδώ πέρα σε γενικές γραμμές. Να πω το εξής. Τι είναι το σημαντικό για εμάς. Και το τι έχει συμφωνηθεί. Το ότι δηλαδή θα πρέπει από τις επόμενες ευρωεκλογές να έχουμε δύο υποψηφίους, έναν άντρα και μία γυναίκα για να μπορέσουμε να επιλέξουμε. Η Κομισιόν θα πρέπει να έχει μία ξεκάθαρη προθεσμία υποβολή... του καταλόγου των υποψηφίων στο Κοινοβούλιο και κάτι άλλο. Μετά την τελευταία ακρόαση ε, ήταν σαφές πως αυτά τα τρία λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας συχνά να πω ότι απλά μπορούσαμε και έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά μια διαδικασία και HDI ή κάτι ανάλογο έτσι ώστε μετά την απάντηση του υποψηφίου επιτρόπου να μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Αλλιώς και το ξέρουμε όλοι το ότι γίνεται, διαλέγει ένα σημείο που τον ενδιαφέρει ο υποψήφιος μιλάει γι' αυτό και πέρασαν τα τρία λεπτά. Οπότε θα πρέπει την επόμενη φορά να μπορούμε να ρωτάμε πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτό το οποίο θέλουμε. Αυτά είναι τα σημαντικότερα. Και βεβαίως ε, Υπάρχει εδώ πέρα και η πρόταση να αλλάξει η κατανομή του χρόνου ομιλία. Αυτό δεν μας ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Θέλουμε να τηρηθεί η αρχή Ντεόντ. Ευχαριστώ. Φώστερ. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την δουλειά που έχετε κάνει. Εμεί συμφωνούμε απόλυτα με την ανάδειξη του αυτού που είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση ό,τι αφορά τα συμβαστικά κείμενα. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε ήδη στο θέμα της ισότητας φύλου. Σε έναν ωραίο κόσμο, πολύ σωστό θα πρέπει να ήταν να έχουμε ισότητα, ισορροπία μεταξύ των φύλων. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε και γι' αυτό είναι σημαντικό η φράση ισορροπία φίλων, να μην πούμε σε πολύ λεπτομέρειε. Γιατί αν ένα κράτο μέλο υποβάλλει υποψήφιο και ο υποψήφιο είναι μια γυναίκα, δεν πρέπει να το δεχθούμε ή όχι λόγω της ε, ικανότητα του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά προηγουμένω θα πρέπει να το κρίνει αυτό το κράτο μέλο. Να υπάρχει λοιπόν μια αναφορά στο ότι πρέπει να υπάρχει σωστή επιλογή των υποψηφίων, προεπιλογή των υποψηφίων. Το λέω αυτό διότι στη δική μα ε, περίπτωση η, η υποψηφιότητα Μπόλτ έγινε πολύ, σε πολύ στενό χρονικό διάστημα και κάποια από τα τεχνικά θέματα είναι δύσκολα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις επιτροπές δεν είναι εύκολο. Πάμε σε πολλές επιτροπές. Η αρχή λοιπόν είναι σωστή, αλλά στη συμβιβαστικό 2 στο αγγλικό κείμενο έχει κάτι σε παχιά και λέει ε, η σωστή έκφραση είναι opposite, take it or leave it. Εν γέννη υποστηρίζουμε το κείμενό σας πάντως με αυτές τις μικρές αλλαγές. Ευχαριστώ. Ο Παβέλ Τελίτσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομος κι εγώ. Πρώτον, πολύ καλό το κείμενο και πολύ καλή και η συζήτηση που είχαμε. Εν γέννη συμφωνούμε με την συμβαστική πρόταση. Τα εξή σημεία εκτιμού. Πρώτον, θα θέλαμε να δούμε τους υποψήφιους να παρέχουν κάποιο πολιτικό πρόγραμμα. Πολλές, ε, πολλοί επιτροποί μας έδωσαν ε, ουσιαστικές προτεραιότητες, πολλές όμως, συγκεκριμένες. Αυτό σε άλλες περιπτώσεις δεν το είχαμε και χαίρομαι που εμφανίζεται αυτό. Για το θέμα της ισότητας φύλων και εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει μια τροπολογία που αναφέρεται στο θέμα της ισότητας φύλων. Θέλουμε ωστόσο δύο υποψήφιους από κάθε κράτος μέλος, διότι η ποιότητα των υποψηφίων είναι πιο σημαντική ακόμα πιο σημαντική, αν μου επιτρέπετε, και από το αν ένα κράτο μέλος δώσει δύο άντρε ή δύο γυναίκε. Είναι σημαντικό λοιπόν και είναι σημαντικό ο πρόεδρο τη Επιτροπής να μπορεί να κάνει επιλογή. Ξέρουμε ότι όταν υπάρχει ένα υποψήφιο σε κάποιε περιπτώσει, ωστόσο, ιδίω δύσκολα μπορεί να αλλάξει την υποψηφιότητα αυτή ο πρόεδρο τη Επιτροπής. Είναι και θέμα πολιτική. Αυτό είναι μια μεγάλη βελτίωση. Το να συμπεριλάβουμε και το θέμα του φίλου, καλό είναι και αυτό. Είχα κάποιες δυσκολίες πρέπει να σας πω με κάποιες από τις τροπολογίες. Να σας τα πω του κ. Βαντερκάμπ. Το σύστημα DON'T. Εμεί μιλάμε για κομισιόν τώρα. Για ένα πολιτικό όργανο. Για μια κυβέρνηση, τέλο πάντων την ε, το πρόσωπο της Ευρώπης. Το να βάζουμε το σύστημα DONT τώρα, ε, πάει πολύ. Παρά είναι σημαντικό εγχείρημα για να μπει στη διαδικασία του συστήματος DONT. Το δεύτερο θέμα για, τη ίδια για την ίδια τοπολογία είναι αυτό το ping-pong. Εμείς τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε όσο πιο διαδραστική γίνεται. Μία ερώτηση, μία απάντηση. Και ενδεχόμενο να επανέλθει κάποιος. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που δεν υποστηρίξαμε, που δεν υποστηρίχθηκαν. Μία αμφιλεγόμενη που το έχω δει ωστόσο είναι κάποιοι επίτροποι σε επιτροπές κατά βάση δεν μπορούν να έρθουν να επικοινωνήσουν με το κοινοβούλιο σε γλώσσα άλλη από τη δική τους. Αυτό είναι για μένα μήνυμα ότι κάποιοι δεν είναι επαρκώς άνετοι σε άλλη γλώσσα πριν τη δική τους. Αυτό είναι ατυχές. Τρεις-τέσσερις επίτροποι απαντώντας δεν μπορούν να κάνουν διάλογο σε άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής τους. Προφανώ δεν πρέπει να γνωρούμε κάτι φυσικό. Ένα Γάλλο, ένα Άγγλο, ένα Γερμανό χρησιμοποιούν τη γλώσσα του, αλλά ένα μελλοντικό Τσέχο ε, υποψήφιο θα ήθελα να μπορεί να απαντήσει σε μια γλώσσα άλλη πέραν των τσέχικων. Αυτά προς το παρόν. Η πρόταση είναι καλή. Θα περάσει. Και αν γίνει δεκτή από την Επιτροπή, θα έχουμε προχωρήσει καλά. Ευχαριστώ Μαρία Κέλεν. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ καλή αυτή η έκθεση. Αυτό που είναι σημαντικό για το μέλλον είναι οπωσδήποτε το ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια να επιτευχθεί μια ισορροπία των φίλων στην Κομισιόν και θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τις ε, ικανότητες ε, και την ισορροπία των φίλων. Και βεβαίως να λάβουμε υπόψη και τις απόψεις των επιτροπών. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω πώς θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το, το θέμα των διαδικασιών των επιτρόπων. Καταρχάς, να τονίσω την ανάγκη να αναφέρονται οι δηλώσεις συμφέροντος των υποψήφιων για να μην φτάνουμε σε ακροάσεις με πλήρη αδιαφάνεια του αν έχουν μετοχές, επιχειρήσεις που είναι ασυμβίβαστες με την εντολή που θα λάβουν αν εκλεγούν. Δεύτερον, για τις γλώσσες, όντως. απαιτείται να ξέρει ένας οποιοδήποτε υπάλληλο μια άλλη γλώσσα. Ε, πρέπει να απαιτείται και από του επιτρόπου. Να λάβουμε υπόψη επίση ότι κάποιοι μπορεί να ξέρουν και γλώσσε μη ευρωπαϊκέ. Καλύτερα να ξέρουν ευρωπαϊκέ δηλαδή. Οπότε και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Για το θέμα τη ισότητα των φίλων. Εγώ θα μιλούσα περισσότερο για θέμα για ίσες ευκαιρίες ανδρών γυναικών. Όλο, αυτό που ακούμε πάντα είναι ότι ωραία να έχουμε ποιότητα καλύτερα να είναι άντρες αν είναι καλοί. Ε, Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών έχει προτείνει για το ελεκτικό συνέδριο να υπάρχει τουλάχιστον ένας και μία υποψήφια από κάθε κράτος μέλος. Να υποχρεώσουμε λοιπόν τα κράτη να υποβάλουν κατελάχιστον υποψηφιότητες ενός άνδρα μιας γυναίκας. Όποιον θέλουν, αλλά να ψάξουν. Γιατί δεν ψάχνουν. Παίρνουν τον δικό τους και τον βάζουμε. Και ξέρουμε ότι έχουν κολλητό περισσότερο από ότι κολλητή. Και αυτούς βάζουν. Να τους βρείτε, να τις βρείτε και να το συζητήσουμε μετά. Κατόπιν. Μήπως ήταν σκόπιμο να μπορούμε να έχουμε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο για τους ε, υποψήφιου επιτροπές, οι επιτροπέ όπως οι δικοί μα που είναι τεχνικέ, το βλέπουμε κιόλα ότι η αλλαγή τη υποψήφια δεν μας επέτρεψε να έχουμε καλή εικόνα των γνώσεών τους. Να έχουμε λοιπόν γραπτές ερωτήσεις που θα τι υπογράφει ο υποψήφιος ή η υποψήφια, Οπότε ώστε να ξέρουμε ότι δεν το ετοιμάζουν μόνο υπηρεσίε και τα λένε, αλλά τέλο πάντων να ε, γιατί ξέρουμε ότι προπονούνται οι υποψήφοι για να έρθουν στις ε, ακροάσεις, αλλά να μπορούν να υπογράψουν, να πρέπει να υπογράψουν τις απαντήσεις τους οι επίτροποι για να δεσμεύονται κατόπιν από αυτές. Λουσί Άντερσον, εγώ συμφωνώ με αυτή την έκθεση, είναι εξαιρετική και είναι καλό το ότι έχουμε συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω πως η διαδικασία αυτή έχει επικριθεί και αλλού, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω πως προσελκύει και την ε, προσοχή της κοινή γνώμης και αυτό είναι κάτι το θετικό και πρέπει να λάβουμε υπόψη και πολύ σοβαρά. Σε κάποιες άλλες επιτροπές νομίζω υπήρχε μια διαδικασία όπου κάποιοι υποψήφοι ε, κλείθησαν ξανά και νομίζω πως πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε αν ε, κάποιος ε, όπως είπα δεν υπερκείς να μπορούμε να τον ξαναφέρουμε πέρα. Για το θέμα της ισορροπίας των φίλων συμφωνώ με την Ινές και, άλλου, και άλλους. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχουν ικανές γυναίκες και αν δεν απαιτηθεί από τα κράτη-μέλη να προτείνουν γυναίκες δεν θα το κάνουν. Δεν δέχομαι ότι δεν υπάρχουν ικανές ε, υποψήφοι. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα και επίσης πρέπει να σημειώσουμε. Εγώ είμαι απογοητευμένη με το σχόλιο της κυρίας Τζάκη Φώστερ γιατί εμείς έχουμε εμπειρία εδώ πέρα και η στάση του κόμματός της είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν περισσότερες γυναίκες ε, ε, βουλευτίνες των εργατικών από ότι όλα τα άλλα κόμματα μαζί. Γιατί εμείς παίρνουμε τέτοια μέτρα. Και να με σαφείς εδώ πέρα. Επιτρέπουν, επιτρέπει θετικές δράσεις το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όχι θετικές διακρίσεις, αλλά ε, να διακρίνουμε εδώ πέρα μεταξύ θετικής δράσης ε, που και θετικής διάκρισης η οποία δεν επιτρέπεται. Οπότε θα πρέπει εδώ πέρα νομίζω να επιμείνουμε σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια και την υποστήριξη. Να πω κάτι τώρα για το θέμα των φίλων. Στη συνθήκη τη συνταγματική που απορρίφθηκε βεβαίως υπήρχε μια πρόβλεψη ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τρεις ε, υποψήφοι, εκ των οποίων τουλάχιστον μία γυναίκα. Και ο Γιούνκερ είχε πει πως ήθελε τουλάχιστον τόσες γυναίκες όσες είχε και η Επιτροπή Μπαρόζο. Παίζει λοιπόν κάποιο ρόλο και δεν ξέρω τώρα να, αν πρέπει να φτάσουμε στο τελευταίο αυτό σημείο να έχουμε ε, να επιλέγουμε αυτό αν είναι άντρα ή γυναίκα, αλλά θα πρέπει κάθε χώρα να προτείνει δύο. Για την διαδικασία και FDI τώρα εδώ πέρα σκεφτήκαμε πώς θα δομηθεί αυτή η διαδικασία. Και τελευταία στιγμή η διάσκεψη των Προέδρων μας είπε θα κάνετε αυτό. Αυτό είναι πρώτον αναξιοπρεπές και η διάσκεψη των Προέδρων δεν πρέπει να ασχολείται με το πώς εμείς στην Επιτροπή θα βρούμε μια συνενετική λύση για το θέμα αυτό και θέλουμε αυτή την ευελιξία. Εμείς δηλαδή ως Επιτροπή να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Με το γραπτό ερωτηματολόγιο η... δεν μ' ακούει η Νέσα Γιάλα Σέντερ. Θα το πω λοιπόν. Το είχαμε στο παρελθόν, τα γράφαν όλα εκεί πέρα και το ξέρω. Ε, απ' έξω ούτως ή άλλως. Τώρα δεν ξέρω ποιος τα γράφει, ποιος γράφει αυτές τις απαντήσεις. Εμένα δεν μ' αρέσουν Κοστίζει χρόνο, κοστίζει χρόνο στους υπαλλήλους που τα γράφουν και σε τελικά κανείς δεν αναφέρεται σε αυτές τις απαντήσεις. Γιατί όλοι σκέφτονται δεν παίζει κανένα ρόλο, σημασία έχει τι θα πούνε εδώ πέρα και να ξαναρωτήσω. Οπότε μπορούμε να γλιτώσουμε χρόνο και χαρτί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη στήριξη. Η ψηφοφορία είναι αύριο στη δική μας την Επιτροπή, 17 Ιουνίου στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και η Ολομέλεια ψηφίζει τον Ιούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σημείο 6. Ολοκληρωμένη πολυτροπική έκδοση εισιτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Dieter Λέμπρεχτ Κοχ. Είναι η της. λοιπόν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, στόχος μου είναι να δούμε την παροχή ολοκληρωμένης πολιτικής έκδοσης εισιτηρίων, πληροφοριών και λοιπόν ταξιδιωτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να έχουμε μια κινητικότητα που θα είναι προσανατολισμένη στον επιβάτη και θα, τον, θα το επιτρέπει να κινείται από πόρτα σε πόρτα. είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ευρωπαϊκή πολιτική συγκοινωνιών, γιατί θα αυξηθεί έτσι η αηφορία και η ενεργειακή ε, αποτελεσματικότητα, θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα αποφύγουμε τα μποτιλιαρίσματα, θα έχουμε κοινωνική κινητικότητα, καλύτερο τουρισμό και θα δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας, καθώς και ε, πέμπτον βεβαίως θα ενισχύσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα γίνει πιο ελκυστική η Ευρώπη. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει οθήσεις για την στρατηγική αυτή. Παρά το ότι έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες για αυτό το ζήτημα, συχνά είναι σε επίπεδο κρατών μελών ή περιφερειών. Και κατά κανόνα σε συγκεκριμένες εταιρείες. Ε, οι πλατφόρμες που υπάρχουν δίνουν πάρα πολύ μικρές δυνατότητες και κατά κανόνα βεβαίω ε, έχουν στηθεί από διάφορα εμπορικά συμφέροντα. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν επαρκεί. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα για ε, μια ίση δίκαιη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ε, πολυτροπικής έκδοσης ε, εισιτηρίων έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να έχει αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες γιατί μόνο τότε θα είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στην, ε, σε αυτό το οποίο θέλει. Ίσως την πιο το πιο γρήγορο ταξίδι, το πιο φτηνό, το πιο αηφόρο. Αναμένουμε λοιπόν εδώ πέρα από την Κομισιόν προτάσεις για μια πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά την έκδοση των εισιτηρίων ή τη μορφή των δεδομένων, η Κομισιόν δεν πρέπει να καθορίσει εδώ πέρα προδιαγραφές. Ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίσεων. Η πολιτική πρέπει να δημιουργεί το πλαίσιο, όχι να δίνει τις τεχνολογικές λύσεις. Άρα η νομοθεσία δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής σε επίπεδα που θα είναι ε, πάρα πολύ υψηλά. όπως είπα θα μπορούσαν ε, οι διάφορες εταιρείες να συμφωνήσουν σε μια πλατφόρμα ε, η οποία βεβαίως μετά θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατανομή των εισπράξεων. Βεβαίως οι εταιρείες δεν θα πρέπει να εμποδίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε αυτό. Το αντίθετο. Πρέπει να τις ενισχύσουμε, να τις βοηθήσουμε μέσω παραδείγματος χάρη διαφορών προγραμμάτων ενίσχυσης. και βεβαίως ε, οι τοπικές ε, συγκοινωνίες ε, παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς είναι το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι και σκέλος κάθε ταξιδιού. Και χωρίς αυτές δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχει κάποιος μια ολοκληρωμένη εικόνα και πρόγραμμα του ταξιδιού. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δημιουργηθούν εθνικά συστήματα προγραμματισμού ταξιδιών και μετά δικτύωσή τους διασυνοριακή. Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο έχουν τεράστια σημασία, ειδικά στην εποχή του smartphone ο ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πριν και κατά τη διάρκεια ενός ε, ταξιδιού να βλέπει και καθυστερήσεις και εναλλακτικέ διαδρομές. Εδώ πέρα το Γκαλιλαίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Τέλος, θα πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικά αυτά τα ταξίδια για... με το να ξεκαθαρίσουμε τα δικαιώματα των επιβατών. Κάτι το οποίο σήμερα είναι ανοιχτό ειδικά σε ε, ζητήματα ευθύνης αστικής. Όπως είπα, στόχος είναι ένα πολυτροπικό ιστήριο, αλλά πρώτα απ' όλα μια δίκαιη και ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο πριν κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μας ε, έχει οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα. Οπότε θέλουμε ήδη πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού να ψηφίσουμε την έκθεση. Οπότε θα πρέπει 4 με 5 Μαΐου να συζητήσουμε τις τροπολογίες στην Επιτροπή μας και μέσα Μαΐου να συναντηθούν οι σκιώδεις εισηγητές και 28 Μαΐου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και μετά να πάμε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο, το αργότερο τον Ιούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η Γιάννης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή ότι είναι πολύ καλό το προσχέδιο τη έκθεση. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτή η ενοποίηση του συστήματο έκθεση πολυτροπικών εισιτηρίων θα έχει πλέον εκτήματα για όλη την Ευρώπη. Ε, υπάρχουν ήδη εξελίξει τι οποίε όμω πρέπει να ενθαρρύνουμε για να επιταχύνουμε γιατί ακόμα οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Ο εισηγητής αναφέρει πολλές από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Τα εξή σημεία είναι σημαντικά κατά την άποψή μου. Ο εισηγητής λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους σε παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ε, που σε ταξιδιωτικά γραφεία, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, να προτείνουν αυτές τις δυνατότητες στους πελάτες τους. Όμως εδώ έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα, γιατί ε, διάφοροι πάροχοι ε, υπηρεσιών προσπαθούν να κατακτήσουν εκείνοι τους καταναλωτές και να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Και ήδη στην Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί ε, στον τομέα του σιδηροδρόμου για παράδειγμα ε, μεγάλα συστήματα τα οποία τα έχουν δημιουργήσει μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείε και οι οποίες συνειδητά έχουν αποκλείσει τις μικρότερες εταιρείε από τις πρόσβαση στα συστήματά τους αυτά. που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πρότυπα ε, πρόσβασης στην αγορά. Για να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Τώρα, για να ε, επιβληθεί κάτι τέτοιο, μπορεί να χρειαστεί η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλειών. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση με ένα άλλο σημείο της, της έκθεσης του εισηγητή, που λέει ότι καλό θα ήταν να αποφύγουμε την νέα νομοθεσία, τη νέα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Πάντως νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια ανοιχτή πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ε, και για να γίνει αυτό λοιπόν απαιτείται νέα νομοθεσία. Άρα ε, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Θα χρειαστούν δεκαετίες εάν ε, επιδιώξουμε να πείσουμε τους, ε, τις διάφορες εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να το κάνουν αυτό εθελοντικά. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί νομοθεσία. Ένα αντιφυστικό πλαίσιο ώστε να αναγκαστούν να το κάνουν. Πάντω, σε γενικέ γραμμέ ε, συμφωνώ με, αρκετά με τη συζήτησή σα και θα την ενισχύσω με τροπολογίε. Τζάκι Φώστα, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Κοχ θα θυμάται και από την προηγούμενη θητεία το είχαμε συζητήσει το ζήτημα ότι ήταν αδύνατον για πολλούς από τους επιβάτες να αγοράσουν ένα εισιτήριο τον οποίο να καλύπτει πολλές διαδρομές σιδηροδρομικές. Δηλαδή ακόμα και μένοντας στον ίδιο τρόπο μεταφοράς, στο ίδιο μεταφορικό μέσο, φανταστείτε τι συμβαίνει στις πολυτροπικές μεταφορές. Εάν κάποιος επιθυμεί να ταξιδέψει την Φιλανδία μέχρι την Ιταλία, θα αναγκαστεί να αγοράσει πολλά διαφορετικά εισιτήρια. Είμαστε λοιπόν πολύ μακριά από μια ιδανική κατάσταση, όμως συνεχίζω να είμαι οπτιμίστρια προσωπικά. Να αισιοδοξώ. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα καλά παραδείγματα. Πριν από 40-50 χρόνια στις αεροπορικές μεταφορές η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Αγόρασε κανεί ένα εφορικό εισιτήριο, δεν γνώριζε σε ποια χώρα θα καταλήξει και σε ποια χώρα θα καταλήξουν οι αποσκευέ του. Αυτό σήμερα έχει αλλάξει τελείω φυσικά. Επομένω έχει υπάρξει πρόοδο στη... στον κλάδο των μεταφορών και καλά παραδείγματα. Θετικά παραδείγματα. <clears throat> Σε ορισμένα κρατημέλη, για παράδειγμα στο Λονδίνο έχουμε μια κάρτα η οποία σας επιτρέπει να κινείστε στο μετρό, στο σιδηρόδρομους και σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια νέα κάρτα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε τις πρακτικές και είναι κέρια η στιγμή που έρχεται η έκθεσή σας. Το ζήτημα λοιπόν είναι με ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα ενισχύσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να προέλθει από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη-μέλη βρίσκονται πιο μπροστά από άλλα στο θέμα αυτό. Και πρέπει να προσέξουμε να μην έρθει από τι Βρυξέλλε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο στην πραγματικότητα να καταπνίξει τι όποιε πρωτοβουλίε ήδη υπάρχουν. Και ένα σημαντικό θέμα είναι τα δικαιώματα των επιβατών, τα οποία τα έχουμε καλύψει με νομοθεσία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα τα ζητήματα ε, που έχουν σχέση με τις θελάσσιες μεταφορές, τι συμβαίνει σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης. Γιατί το λέω αυτό, φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για πολλά μεταφορικά μέσα που πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους. Εάν έχουμε να πάρουμε ένα φεριμπότ για να φτάσουμε στο αεροδρόμιο, για να πάρουμε ένα αεροπλάνο να φτάσουμε στο τρένο, ποιος θα πληρώσει σε περίπτωση καθυστέρησης που διακόψει αυτή τη συνεχή μετακίνηση πρέπει να προβληματιστούμε για το ποιο είναι το καταλληλότερο νομοθετικό πλαίσιο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Πάντως πιστεύω ότι η έκθεσή σας είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Και είναι ένας τρόπος να βάλουμε προθεσμίε έτσι ώστε να κοινοτοποιήσουμε τα διάφορα κράτη-μέλη και να, να, να αρχίσει να συζητάτε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Παύλ Τελετσικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κοχ και για την πρωτοβουλία και για το κείμενο δύσκολο και μεγάλο θέμα. Το πρώτο ερώτημα που έχετε στο μυαλό μου είναι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπρος έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν μια σειρά έργων που λειτουργούν σε κάποια κρατημέρη ακόμα και διασυνοριακά ή θα το δούμε μόνο από την οπτική της εσωτερικής αγοράς. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να δούμε πού είναι τα προβλήματα, πώς τα αντιμετωπίζουμε, αν χρειάζεται ένα κανονιστικό, νέο κανονιστικό πλαίσιο, η χρηματοδότηση πιθανή. Ε, αν μιλάμε για διασυνοριακό στα περιφερειακά τρένα, ε, η κατάσταση είναι απλούστερη. Πρόκειται λοιπόν για δύο διαφορετικές ε, περιπτώσεις. Τώρα, για τη φιλοδοξία μας. Υπάρχουν όντως δυσκολίες, τα bottlenecks, και απλά πρέπει να, και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι, ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες. Εγώ υπέβαλα κάποιες τροπολογίες για να δείξω ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα ακόμα στενοπή σε σχέση με αυτές που εντοπίζει το κείμενο. Μιλάμε για ασύμβατότητα προτύπων, μηχανογράφησης, τι εννοούμε πλατφόρμα. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Μερικές φορές μιλάμε για πραγματική πλατφόρμα, ένα τυποποιημένο σύστημα ε, και κάτι τέτοιο σημαίνει τεράστιο κόστος και αυτό με ξαναφέρνει στο θέμα του πόσο φιλόδοξοι είμαστε. Να μια στενοπός λοιπόν. Οι άλλοι που αφορά ένα θέμα που το συζητάμε στο και καιρό είναι ότι δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο λειτουργίες μεταξύ όλων. Δύσκολο μπορούμε να έχουμε ε, ένα ενοποιημένο σύστημα έκδοση εισιτηρίων αν δεν υπάρχει ισότιμη, ε, ισότιμο πεδίο για όλους. Και αυτό είναι ένα θέμα κινήτρων εν πωλής. Μετά, το σύστημα, το εισιτήριο ενσωματώνεται στο σύστημα έκδοση εισιτηρίων, δηλαδή ένα εισιτήριο θα είναι ή πολλά διαλειτουργικά ενοποιημένο ή συνδεδεμένο σύστημα. Θα πηγαίναμε μέχρι το να φτάσουμε σε μια σειρά εμποδικών ρυθμίσεων μεταξύ των φορέων και μετά μπαίνει το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών. Ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικά δικαιώματα επιβατών στις ιδεοδομικές και διαφορετικές αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά θεμάτων. Προφανώς κάποια από τα προβλήματα αντιμετωπίζονται, πρέπει να αντιμετωπιστούν νομοθετικά, αλλά όχι. Υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης. Εγώ θα ήθελα ένα πλήρως ενοποιημένο σύστημα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό. Λάβετε επίσης υπόψη και αυτό που συζητήσαμε πριν λίγο. Έύσα μια ευκαιρία. Το ταμείο δηλαδή. Ε, το ταμείο Γιούνκερ πού αλλού θα μπορούσε να δουλέψει καλύτερα από ότι σε κάποια τέτοια καινοτόμα δράση. Θα σταματήσω εδώ. Πρόκειται για, μια, για ένα κείμενο που αποτελεί πολύ σωστή στέρεη βάση από πλευράς φιλελευθέρων θα υποβάλω μια σειρά ε, τροπολογιών που ενδεχομένως να δείχνουν και τις πιθανές λύσεις. Αλλά είναι κρίσιμο να ξέρουμε πόσο φιλόδοξοι θέλουμε να είμαστε. Ενιαία αγορά, περιφερειακές αγορές. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρία Κελίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Πολύ σημαντική η συζήτηση. Πρέπει να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι τώρα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου του τουρισμού στην Ευρώπη. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει την πρόθεση πολλών πολιτικών και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα αυτό και να βρούμε και τρόπους επιτάχυνσης της διαδικασίας. και πιστεύω ότι μια καλή λύση στον τομέα αυτό θα είναι μια καλή λύση για την Ευρώπη. Στο ε, euh, Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου που δεν μπόρεσε να παραστεί το προσώπο. πω λοιπόν του οικολόγου. Θέλω να σα ευχαριστήσω για το έργο σα. Με την έκθεσή σας αναδεικνύεται πολλά θέματα που οι οικολόγοι τα θεωρούν πολύ σημαντικά και γι' αυτό ίσως ορισμένα, σε ορισμένα από αυτά θα θέλαμε να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος, σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων, είναι ένα ζήτημα ευαίσθητο, γιατί συνδέεται άμεσα με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και ταυτόχρονα θα έπρεπε πιστεύω να επαναξετάσουμε τα διάφορα προγράμματα που ήδη συγχρηματοδοτεί και ήδη ε, εξελίσσονται μέσω της έκθεσης για την ενοποίηση την οποία έχετε επισυνάψει ως παράπτυμα στην έκθεσή σας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε αυτά τα διάφορα project και να δούμε αν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που μπορούμε να λύσουμε από αυτές. Ευχαριστώ, Λούση Άντερσον. Ευχαριστώ. Η εκθέση αυτή είναι πολύ σημαντική και συνδέεται άμεσα με το υπόλοιπο έργο της Επιτροπής μας. Για παράδειγμα την εκθέση στην οποία συνεργαζόμαστε με τη συνάδελφο Καριμπέλη. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες προτάσεις την έκθεσή σας, τις οποίες θα ήθελα να καλωσορίσω, ιδιαίτερα το άρθρο 11, που αναφέρεται στα άτομα με ε, αναπηρία και τα άτομα με κινητικούς περιορισμούς. Περιορισμένη κινητικότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προσπαθήσαμε να αναδείξουμε στην Επιτροπή το προηγούμενο Σεπτέμβριο. Γιατί στις περισσότερες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εταιρείες δεν δίνεται η δυνατότητα σε άτομα που χρησιμοποιούν ε, ανεπιρκές καρέκλες να κλείνουν θέση των προτέρων ε, που θα τους εξασφαλίζει την προσβασιμότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, γνωρίζω ότι έχει συζητηθεί το θέμα των τελών, ε, των ε, συνδρομών πιστωτικές κάρτες κτλ. Πρέπει να εξετάσουμε και το ζήτημα των μεθόδων πληρωμής. Έχει μεγάλη διαφορά εάν κανείς θα δίνει τη δυνατότητα ε, εξόφλησης του τιμή του εισιτηρίου μέσω PayPal ή ποια θα είναι ε, το επιπλέον κόστος το οποίο μετακυλείται στον επιβάτη ανάλογα με, το μέθοδο, με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγει. Γιατί πολλέ φορές Επίσης κάτι άλλο είναι το, το, εμπορικό τα εμπορικά μυστικά τα οποία πολύ συχνά τα χρησιμοποιούν ως δικαιολογία οι εταιρείε για να μην μας δίνουν πληροφορίες τις οποίες ε, είναι προς το δημόσιο συμφέρον είναι διαθέσιμες και θα βελτίωναν και την, ε, τις που παρέχονται στους επιβάτες. Μια και διαφώνησα με την Τζάκη, θέλω να την ευχαριστώ που ανέφερε το ζήτημα του Λονδίνου και τι ενιαίε κάρτε μεταφορά. Παρόλο που δεν συμφωνώ σε τι υπόλοιπε θέσει τη όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν θα πρέπει να υπάρχει για την επικίνδυνο κτλ. Αλλά πράγματι συμφωνώ ότι υπάρχουν πρωτοβουλίε και πρέπει αυτό να φαίνεται στην έκθεση. Στο Όλγα Σελένοβα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάποιες ε, ιδέες. Χαίρομαι που μιλάμε για τα δικαιώματα των επιβατών και το περίπλοκο ζήτημα της χρηματοδότησης γιατί κάποια έργα αφορούν την ολοκληρωμένη αγορά των εισιτηρίων και έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρέπει να τα συμπεριλάβουμε εδώ πέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Νίλσεν ε, για το ζήτημα της ε, πληροφόρησης ε, και το ότι θα πρέπει οι εταιρείε να να συμμορφώνονται με κάποιους κανόνες. Αυτό είναι βασικό ζήτημα της όλης υπόθεσης. Χαίρομαι που αναφέρετε τα άτομα με αναπηρία και ειδικά προβλήματα κινητικότητας και να αναφέρω και τον πληθυσμό ο οποίος γυράσκει και υποτίθεται ότι θα μας απασχολεί στο μέλλον και οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία όλα αυτά. Αλλά δεν πρέπει να δημιουργούμε νέα εμπόδια σε ομάδες πολιτών στο μέλλον. Τέλος. Όταν μιλάμε για ψηφιακή εσωτερική αγορά, μιλάμε και για θέσεις εργασίας ε, και πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα κατά νου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ισμαήλ Ερτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δουλειά που έγινε από εισηγητή και σκιώδης εισηγητές. Θυμάμαι πως το είχαμε αυτό το πράγμα την τελευταία περίοδο και αν ε, δεν κάνω λάθος το ίδιο πράγμα είχαν πει τότε. Πώς θα καταφέρει ο απλός πολίτης να έχει τόσες πληροφορίες στη διάθεσή του ώστε να μπορεί μετά να κανονίζει μόνος του το ταξίδι του. Και νομίζω πως πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό τον στόχο και να τον ακολουθήσουμε προσιλωμένα. Τώρα, η αγορά, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη κάποιες προτάσεις, λύσεις. Βεβαίω, ε, αν ο καθένας ε, κάνει το δικό του είναι κατακαιρματισμένα και δεν ε, συνδέονται. Και να πω πως εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω και μίλησα και με κάποιους ανθρώπους να παραμείνει αυτό στο χέρι των επιχειρήσεων. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω τώρα πραγματικά να ε, κάνουμε εμείς την δουλειά κάποιων άλλων. Ε, τώρα δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά βλέπετε πως ε, οι μηχανές αναζήτησης ήδη υποκαθιστούν ε, τις εταιρείες ε, ταξιδιών και θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια αυτών των επιχειρήσεων και πρώτα απ' όλα σε επίπεδο εθνικό και μετά από μια μεταβατική περίοδο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρξει αυτή η δικτύωση δηλαδή. Και το ε, λέω και θα το ξαναπώ. Δεν πρέπει να φτάσουμε μέχρι του σημείου μετά οι εταιρείε ε, να πρέπει να δημοσιεύουν ε, εμπορικά μυστικά. να έχουμε τις φλοφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής και υπάρχουν ήδη σε μηχανές αναζήτησης στον τομέα των αερομεταφορών πατάμε και βλέπουμε ποια εταιρεία προσφέρει ποια δρομολόγια, τι ώρα. Χωρίς όμως αυτό να ε, υποχρεώνει τις εταιρείες μας να φανερώνουν εμπορικά μυστικά, το πώς υπολογίζουν τις τιμές κτλ. Και μετά να το εκμεταλλευτούν άλλες ε, εξωευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ε, είναι αυτό που συζητούμε είναι πολύ σημαντικό θέμα. Σύμφωνο ότι ένα καθοριστικό θέμα είναι το, δρομο, το δρομολόγιο και τα ωράρια όταν προετοιμάζεις ένα ταξίδι. Το άλλο είναι η αγορά των εισιτηρίων, η πόλη των εισιτηρίων. Θα θέλω λοιπόν να ξέρω περισσότερα στην έκθεση για το εξή. Οι δύο αυτές παράμετροι πρέπει να είναι λεπτομερέστερες, να ορίζονται καλύτερα. Εμείς όταν μιλούμε για δρομολόγια. Το είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Υπάρχουν επιχειρήσεις σε παγκόσμιο, εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θέλω να πω ονόματα, που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Μπορείς να φτιάξεις ένα δρομολόγιο με αυτοκίνητο, με ποδήλατο, με περπάτημα, με δημόσιες μεταφορές, χωρίς πρόβλημα. Άρα, ο προγραμματισμός ενός δρομολογίου, μιας διαδρομής, είναι εφικτός. Αυτό που είναι πιο ευαίσθητο είναι το θέμα της πώληση, της έκδοσης και πώληση των εισιτήριων για τη συγκεκριμένη διαδρομή. υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μονοπόλιο σε μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να μην υπάρξει τέτοια, τέτοιο μονοπόλιο. Ε, άλλο θέμα είναι αν είναι αναγκαίο ή ρεαλιστικό να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα έκδοση εισιτηρίων στις παλιές, σε παλιότερες συζητήσεις στο παρελθόν είχαμε ήδη αναφέρει ότι μπορούμε να αναμένουμε συγκρούσεις ή διαφορές μεταξύ των συμφερόντων που έχουν τα διάφορα είδη μεταφοράς. Ένα ενιαίο σύστημα έκδοση εισιτηρίων θα έχει μια σειρά ζητημάτων. Καλό είναι που ξεκινούμε να το συζητούμε το θέμα αυτό, αλλά και πάλι πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, μάλλον θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για το θέμα αυτό από ό,τι νομίζουμε. Ωραίο είναι το ότι ο εισηγητής μιλά για τα άτομα με αναπηρίες. Αγνοείται εν το ζήτημα αυτό. Ιδίως σε κάποια από τα λιγότερα ανεπτυγμένα κράτη-μέλη σε επίπεδο υποδομών βεβαίως, που πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Θυμάμαι στο τρίτο συνδρομικό πακέτο πριν από 8-9 χρόνια λέγαμε πως θα πρέπει να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες ε, διαθέσιμες πανευρωπαϊκά και το ίδιο με τα ειστήρια. Και δοκίμασα, δηλαδή μπορώ να βγάλω ένα ειστήριο Βρυξέλλες ε, Κολονία αλλά μετά Βρυξέλλες Μίχελστατ ε, δεν γίνεται. Εντάξει, είναι ωραία τα εμπορικά μυστικά, αλλά οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν τα ίδια προβλήματα. Ούτε αυτέ θέλουν να δίνουν πληροφορίε. Αλλά λειτουργεί το σύστημα. Γι' αυτό θεωρώ πως το εμπορικό μυστικό είναι δικαιολογία που τελικά την πληρώνει ο πελάτης για να διατηρήσουν το μονοπωλιό τους. Γιατί οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ούτε μία σχέση με εμπορικά μυστικά. Θέμα να ξέρουμε πότε πηγαίνει ποιο τρένο πού. Ούτε αυτό δεν μας λένε. Και η Κομισιόν κάτι πρέπει να κάνει. Δεν έχω δει καμία διαδικασία να κινηθεί ε, να κινηθεί διαδικασία κατά εταιριών που δεν δίνουν τις πληροφορίες. κάθε κανείς δηλαδή στην αποβάθρα και εμφανίζεται η πληροφορία όταν έρχεται το τρένο το ίδιο. Ποιο τρένο είναι. Γιατί δεν θέλουν να, να φανερώσουν τις πληροφορίες οι εταιρείε. Τι να πω, σε κάποιες ε, εταιρείε υπάρχει το 95% των πληροφοριών, σε άλλες 80%. Μα άμα δεν καταλάβουν οι εταιρείε πως είναι προς το συμφέρον τους, κατ' ουσίαν λένε είμαστε η λύση. Πάρτε το κτέλι ή το αεροπλάνο. Έτσι. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Και αν δεν δίνουν τις πληροφορίες, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το είχαμε αποφασίσει ήδη στο τρίτο στερεοδομικό πακέτο. Γιατί δεν κάνει τίποτα η Κομισιόν. Έχετε τον λόγο και περιμένω να ακούσω. Γιατί, Γιατί τότε θα ε, το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δεν θα χρειαζόμασταν την έκθεση. Εάν τα παίρναμε σοβαρά αυτά που λέμε. Η ευθύνη τώρα για την κάθε επιχείρηση τη βελγική, τη γαλλική, τη γερμανική. Είναι σαφές πως έχουν την ευθύνη για διάμορφωση των τιμών. Αλλά τις πληροφορίε θέμε. Αυτό είναι για τον πελάτη. Αν δεν ξέρει ο πελάτης ε, πότε φεύγει το τρένο δεν το χρησιμοποιεί. Και άμα δεν το χρησιμοποιεί μετά κόβεται το δρομολόγιο και το βλέπουμε. Κόβονται δρομολόγια με γεμάτα τρένα. Οπότε μιλάμε για πραγματικά κάτι το οποίο είναι ε, εκ των όν ουκάνευ. Ε, είναι απολύτως απαραίτητο. Πρέπει να μπουν όλα αυτά μαζί σε ένα σύστημα και δεν χρειάζεται να πηγαίνω σε 6-7 site για να βρω τις ε, πληροφορίες για να βγάλω εισιτήρια. Γίνεται με τη μία στις αεροπορικές μπορώ να βρω τα πάντα παντού στον κόσμο και δεν γίνεται στο τρένο. Αυτές τις πληροφορίες τις θέμε, δρομολόγια και τιμές. Λοιπόν, το λόγο έχει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω, με την Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτα απ' όλα. Να σχολιάσω αυτά που είπατε τώρα στο τέλος κύριε Πρόεδρε ότι πράγματι δεν είναι καινούριο το πρόβλημα. Ωστόσο όμως αυτό που έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό είναι να δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και έτσι να αυξάνονται οι προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όπως είπαν και πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου, έχουν υπάρξει μεγάλες εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις και πρόοδος ε, σε ορισμένα μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα ίσως σε ορισμένες περιοχές ή χώρες της Ευρώπης. Αυτό όμως που λείπει είναι η παροχή πολυτροπικών πληροφοριών στους ταξιδιώτες, που δηλαδή θα έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέγουν, να έχουν τις πληροφορίες στη διάθεσή τους για να επιλέξουν ποιο μέσο μεταφοράς ε, θα χρησιμοποιήσουν. Εκεί πάσχουμε. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση ΚΟΧ και ε, μας χαροποιεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της πολυτροπικής ε, μεταφοράς στην Ευρώπη. Ένα θέμα που θα το θυμάστε και από τις συζητήσεις με την Επίτροπο Γκούλτς, ε, που την απασχολεί και εκείνη πολύ και θέλει να το προωθήσει. Ο κλάδος των μεταφορών ε, υφίσταται πολλές αλλαγές και το ζήτημα της πρόσβασης της πληροφορίας έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα γιατί αλλάζει τις επιλογές και τις συνήθειες των ταξιδιωτών. Και οι προσδοκίες λοιπόν των πολιτών μεταβάλλονται και οι συνήθειές τους. Τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο ε, της για τις πολυτροπικές μεταφορές στην Ευρώπη Καλωσορίζουμε λοιπόν για την έκθεση αυτή, γιατί θέματα που αναφέρετε στην έκθεσή σας θα είχαμε αναφέρει και εμείς στο roadmap, στο σχέδιο δράσης. Κάναμε μια, ένα απολογισμό και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάνω από 100 ε, γραφεία ή ε, υπηρεσίες τα οποία ε, δίνουν τη δυνατότητα πολυτροπικής μεταφοράς είτε από ιδιωτικές εταιρείες είτε από εξιδιωτικά γραφεία Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια δυναμική αγορά στον τομέα αυτών που θα έπρεπε να την αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχουν εμπόδια, ιδίω όταν μιλούμε για διασυνοριακές πολυτροπικέ μεταφορές. Τι θα χρειαζόταν για να δημιουργηθούν τέτοιες υπηρεσίες. Το σημαντικότερο είναι προφανές είναι ε, να είναι διαθέσιμα ε, υψηλής ποιότητας δεδομένα ε, τα οποία να είναι και διαλειτουργικά να μπορούν να διαθέσουν μεταξύ τους. Και αν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, αν υφίστανται αυτά τα δεδομένα, μετά μπορούν να χτιστούν οι υπηρεσίες που θα τα αξιοποιούν. Αυτό που πιστεύω είναι σημαντικό να τονίσει το Κοινοβούλιο είναι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα στο θέμα αυτό. Για παράδειγμα, τα ωράρια που είναι ένα θέμα που φυγει η έκθεση. Τα, τα ωράρια τα οποία ανακαλύπτουν μεγαλύτερε μεγαλύτερε μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι και το μόνο που χρειάζεται για να προετοιμάσει κανεί αποτελεσματικά ένα ταξίδι. Υπάρχουν και άλλε μέθοδοι μεταφορά. Για παράδειγμα, ε, το, να ε, μοιραστεί κανεί το κίνητό του με κάποιον άλλον επιβάτη ή το ποδήλατο ή υπηρεσίε οι οποίε απευθύνονται ειδικά σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Και αυτέ οι πληροφορίε θα πρέπει να προσθεθούν. Και πρέπει να δούμε πώ θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα συνθέτει όλε αυτέ τι πληροφορίε και θα τι δίνει ε, προ χρήση κάθε ενδιαφερόμενο. Από την πλευρά μα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζουμε ένα σχέδιο ε, για την πρόσβαση στα δεδομένα για τις πολυτροπικές μεταφορές, με το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα εξή να υπάρχει σεβασμός του ανταγωνισμού και να είναι ξεκάθαρη, να είναι ξεκάθαρη η όρη χρήσης αυτών των δεδομένων. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία για να μην υπάρχει ε, ανισότητα στους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών ε, μέσων μεταφοράς και μεταξύ των διαφορετικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο κάθε τομέα. Δηλαδή να μην δημιουργήσουμε ε, μονοπόλια σε αυτή τη διανομή πληροφοριών Όπως αναφέρει και ο κύριος Κόχ στην έκθεσή του, χρειάζεται η παροχή λοιπόν αυτών, η πρόσβαση σε αυτά τα υψηλή ποιότητα ε, δεδομένα και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και πέρα από το πρώτο βήμα είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία και για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των επιβατών. Το συζητούμε εδώ και πολύ καιρό το ζήτημα των δικαιωμάτων των επιβατών ε, σε ένα ενοποιημένο σύστημα, αλλά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν σκοπεύει εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει η ίδια το σύστημα ε, ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων. Αντιθέτως, εμείς αυτό που θέλαμε να φτιάξουμε είναι ένα πλαίσιο ρυθμιστικό νομοθετικό μας στο οποίο ε, ιδιώτες θα δημιουργήσουν αυτά τα συστήματα. Προετοιμάζουμε, προετοιμάζονται διάφορες πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, ε, η Ένωση Always Traveling ε, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πληροφοριακό σύστημα για την ε, ανταλλαγή ταξιδιωτικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει και την υποστήριξη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Κλείνω λοιπόν μιλώντας για το ζήτημα αυτό των δικαιωμάτων των επιβατών. Συμφωνούμε με τη θέση του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει έλλειψη στην παροχή πληροφοριών στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί για να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις μεταφορές, ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς που θέλουν να επιλέξουν. Επίση, το ζήτημα του ενιαίου εισιτηρίου, σε περίπτωση ενό ενιαίου εισιτηρίου, πρέπει να ρυθμιστεί και, όπως το είπατε εσεί, είναι από το πιο δύσκολα και πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εάν θέλουμε να υπάρχουμε ε, ενιαία εισιτηρία, το ζήτημα τη αστική ευθύνη για κάθε μέρο του ταξιδιού. Και προετοιμάζουμε κάποιο σχέδιο ε, κειμένου και γι' αυτό, Κάποιε ιδέε και γι' αυτό το θέμα. Και τέλος, στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, κάποια από τα θέματα που έθιξαν μέλη της Επιτροπής σας, όπως για παράδειγμα η διαλειτουργικότητα, η πρόσβαση στα δεδομένα ή η πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, διασυνοριακού χαρακτήρα, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μέσω ε, της στρατηγικής αυτής προσβαση σε υπηρεσιες διασυνοριακου χαρακτηρα ολα αυτα ειναι θεματα τα οποια μεσω της στρατηγικης αυτης της επιτροπη θα αντιμετωπίσει. Ευχαριστώ, ο εισηγητής και πάλι. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν είναι πράγματι παλιά ιστορία. Θυμάμαι τη Λευκή Βίβλο 2011, ε, τι γράφαμε εκεί πέρα. Ελπίζω να γίνει κάτι σιγά σιγά. Βεβαίω λόγω του περιορισμού δεν ε, έβαλα κάποια πράγματα στην έκθεσή μου. Τα αναφέρατε εσείς και χαίρομαι ιδιαίτερα για τις τροπολογίες που είναι πάρα πολύ θετικές. Βεβαίω το θέμα είναι προδιαγραφές, ποια δεδομένα, σε ποια μορφή, για να μην έχουμε αφενός μονοπόλια και αφετέρου να έχουν οι επιχειρήσεις την ευκαιρία να ανταγωνίζονται. κυρία Φώστερ και άλλοι ανέφεραν τα παραδείγματα που υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο, διασυνοριακό, τίποτα ακόμα. Αυτή είναι η φιλοδοξία που έχω. Να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια εσωτερική αγορά. Για να δω λίγο. Νομίζω αυτά ήταν τα ουσιαστικά. Νομίζω πως ε, συμφωνούμε με τη λογική της Κομισιόν. Ελπίζω να πάρετε σοβαρά αυτά τα οποία θα πούμε λοιπόν και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα ε, θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους ε, συμμετείχαν, ε, τον εισηγητή, τροπολογίες μέχρι τις 16 Απριλίου, 7 το απόγευμα, 28 Μαΐου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και Ιούλιο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους και κλεισμένων των θυρών. Μόνο τα μέλη της Επιτροπής μας. Μην το παίρνετε προσωπικά. Αυτό θα πει και κλεισμένο των θυρών.